σε δεύτερη ανάγνωση του κυρίου Κονσεγρούα για τη συνεργασία των κατασταλτικών υπηρεσιών. Να μιλήσουμε για την Ευρωπόλ καλύτερα λοιπόν. Κύριε Διέστε Μέρα, έχετε τον λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Και θα ήθελα να καλημερίσω και τον Επίτροπο και όλους τους φίλους που βρίσκονται εδώ. Ε, στον κανονισμό αυτό πρέπει να σας πω πως με έχει απασχολήσει εδώ και τρία χρόνια και πάντα η πρόθεσή μας ήταν η Ευρωπόλ να έχει ένα κανονισμό που θα της δώσει τα παρήτα εργαλεία έτσι ώστε με αποτελεσματικό τρόπο να μπορεί να εκπληρώσει την αποστολή της. Έχει ως βασικό στόχο η Ευρωπόλ να ενισχύσει τις διοκτικές αρχές των κρατών μελών και να υπάρχει αμοιβαία συνεργασία στην πρόληψη και στην καταπολέμηση της τρομοκρατίας, του οργανωμένου εγκλήματος και άλλα 30 εγκλήματα τα οποία έχουν ε, περιγραφεί, για παράδειγμα, οι απαγωγές, οι ομοιρίες, ο ρατσισμός, η ξενοφοβία, οι εκβιασμοί, η παραχάραξη ε, των οικονομικών μεσών, το λαθρεμπόριο ναρκωτικών, όπλων, τη σεξουαλική εκμετάλλευση και έτσι υπάρχουν τέτοια 30 εγκλήματα. Στην ανάγνωση ε, καταφέραμε την πρώτη να αποφύγουμε την συγχώνευση της Europol με τη Σίπολ και πρέπει να σου πω πως το αποτέλεσμα αυτό το πετύχαμε χάρη και στη καλή συνεργασία που είχαμε με τους σκιώδεις εισηγητές για τους οποίους αυτή τη στιγμή θα ήθελα να εκφράσω τις ε, ευχαριστίες μου. Στη δεύτερη ανάγνωση και πάλι είχαμε ένα πολύ υψηλό βαθμό συνεργασίας με τους συναδέλφους και γι' αυτό θα ήθελα να επαναλάβω τις ευχαριστίες μου για τις προσπάθειες που έκαναν αυτά τα τρία μακριά χρόνια των διαπραγματεύσεων. Είχαμε τρεις τριμερείς διαλόγους στην Ιταλική, ε, τρεις στην Λετωνική και τέσσερις υπό τη Λεξοβοργινή Προεδρία και στις 27 Νοεμβρίου πετύχαμε μια καλή συμφωνία και θα ήθελα να σας ευχαριστήσω όλους. Θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω την καταπληκτική δουλειά που έκανε η Βικτόρια Ανταμίτση, η εκπρόσωπος Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τον πολύ ψηλό βαθμό επαγγελματισμού που ε, επέδειξη. Η Ευρωπόλ θα μας βοηθήσει να καταπολεμήσουμε την τζιχαντιστική απειλή. Γι' αυτό λοιπόν θα πρέπει να πρικοδοτηθεί με τα κατάλληλα εργαλεία. Και το ECTC δημιουργήθηκε τον Ιανουάριο, είναι εκείνη η υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης που θα καταπολεμήσει την τρομοκρατία μέσω της ανταλλαγής υπηρεσιών και άλλων καθηκόντων που έχει αναβάλει. Επίσης ε, θα δώσει και νομική βάση στην μονάδα ελέγχου του ε, περιεχομένου του διαδικτύου έτσι ώστε να δούμε ε, το διαδίκτυο τι γίνεται με τις απειλές που εκφράζονται ε, διαδικτυακά έτσι ώστε να μπορούμε να ερχόμαστε σε επαφή με τους παρόχους υπηρεσιών στο ίντερνετ και να μπορούμε και να αποσύρουμε το περιεχόμενο αυτό από το διαδίκτυο αλλά και να εντοπίσουμε αυτούς που κρύβονται πίσω από αυτές τις διευθύνσεις. Θα ήθελα να σας πω πως εδώ στο κείμενο που έχουμε πετύχει είναι μια ανταλλαγή πληροφοριών που θα επιτρέπει και την ανταλλαγή πληροφοριών για εγκλήματα τα οποία θα αναλυθούν και σε επιχειρησιακό επίπεδο και σε επίπεδο ε, νομικό και θα βοηθήσει αυτό και τις διοκτικές αρχές των εθνικών αρχών αλλά όπως επίσης και τους αξιωματικούς συνδέσμους που είναι το σημείο επαφής μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και κρατών μελών. Οι, οι σύνδεσμοι αυτοί θα είναι οι, αυτοί οι οποίοι θα λαμβάνουν αμέσως την πληροφόρηση για τέτοιου είδους αγκλήματα που διαπράττονται. Η Ευρωπόλ με τον τρόπο αυτό θα μπορεί να συνεργάζεται, να συντονίζει ε, κάποιες επιχειρήσεις έτσι ώστε να στηρίζει και να ενισχύει λέξεις κλειδιά τη δράση των κρατώμελων Για πρώτη φορά θα μπορεί να επεξεργάζεται και δεδομένα από ιδιωτικέ πηγές με ένα υψηλό βαθμό προστασίας έτσι ώστε να καταπολεμήσει καλύτερα εγκλήματα τόσο φρικτά όσο η κακοποίηση ανηλίκων. Στα πλαίσια μιας σφριγγυλή αρχιτεκτονικής που θα προστατεύει τα προσωπικά δεδομένα, στα πλαίσια της εποπτείας από τον επόπτη, τον Ευρωπαίο επόπτη, που ως ανεξάρτητο όργανο πάντα θα συνεργάζεται με τις Εθνικές Αρχές Προστασίας Δεδομένων και πάντα θα δεχθεί και μια ιδιαίτερη επεξεργασία και προσοχή στα ευαίσθητα δεδομένα στα πλαίσια του πακέτου που εγκρίναμε την περασμένη Ολομέλεια. Έτσι λοιπόν θα έχουμε μια καλύτερη διακυβέρνηση αυτής της υπηρεσίας, κυρίως μέσω ε, του Συμβουλίου, έτσι ώστε να υπάρχει ένα προηγούμενο για τις υπόλοιπες ε, υπηρεσίες που υπόκεινται σε κοινοβουλευτικό έλεγχο. Στο άρθρο 88 σαφώς λέει πως θα πρέπει να ελέγχονται από τα Εθνικά Κοινοβούλια και από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο οι δράσεις της Europol. Έτσι λοιπόν έχουμε δημιουργήσει μια ε, ομάδα ελέγχου έτσι ώστε η καταπολέμηση του οργανωμένου κλίματος να γίνεται μέσω της καλύτερης δυνατής συνεργασίας μεταξύ των εθνικών αρχών έτσι ώστε και η Eurojust να έχει πρόσβαση στα δεδομένα της Europol. Περάσαμε μια μακρά διαδικασία όμως το αποτέλεσμα είναι καλό και η εργασία ε, θα επιτρέψει στη Europol να εργάζεται 24 ώρες το 24ωρο κάθε μέρα της εβδομάδας. Τίποτα άλλο σας ευχαριστώ κύριε, κυρία Πρόεδρε και κύριε Επίτροπε. Ευχαριστώ. Θα περάσουμε τώρα στον Επίτροπο κύριο Αβραμόπουλο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Αγαπητά μέλη του Κοινοβουλίου, να ξεκινήσω ευχαριστώντας τον εισηγητή μας, τον κύριο Ντία Δεμέρα και την ομάδα του. Έκαναν μια εξαιρετική δουλειά έτσι ώστε να προωθηθεί αυτή η πολύ σημαντική νομοθετική πρόταση. Μετά από τρία χρόνια εντατικής δουλειάς για να καταλήξουμε στη συμβιβαστική πρόταση, τον συγχαίρω για το αποτέλεσμα και τον ευχαριστώ για το πνεύμα συνεργασίας που επέδειξε τι καθιστά τον, κανονικό, τον κανονισμό αυτό σημαντικό. Το θέμα αυτό βρίσκεται καταρχάς στην επικαιρότητα σήμερα, στην κορυφή της επικαιρότητα. Το 82% των πολιτών της Ευρώπης μας λέγουν σε μια πρόσφατη δημοσκόπηση ότι επιθυμούν η Ευρωπαϊκή Ένωση να παρεμβαίνει περισσότερο στα θέματα της τρομοκρατίας από ό,τι το κάνει σήμερα. Αυτή τη στιγμή εφαρμοστεί ο κανονισμός αυτός, την άνοιξη του 17 δηλαδή, θα μας δώσει το κατάλληλο πλαίσιο έτσι ώστε να συμβεί αυτό. Καταρχάς θα καταστήσουμε την Ευρωπόλ κέντρο συλλογή και διανομής πληροφοριών για το σύνολο της Ένωσης. Το Παρίσι και οι Βρυξέλλες μας έδειξαν ποιο είναι το πρόβλημα ξεκάθαρα. Η ανταλλαγή πληροφοριών είναι η αχίλιος πτέρνα μας. Τα κράτη-μέλη θα πρέπει να συντονίζονται στενότερα και αποτελεσματικότερα. Περίπλοκες έρευνες και ανακρίσεις θα πρέπει να υποστηρίζονται από σαφή αναλυτικά στοιχεία. Η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία, η Europol δηλαδή, μπορεί να συνεισφέρει προς την κατεύθυνση αυτή. Και αυτό φυσικά να ελέγχεται δημοκρατικά από το κοινοβούλιο σας οι νέοι κανόνες θα διασφαλίσουν την ανάληψη αυτή ευθύνη σε συνεργασία με τα κοινοβούλια των κρατών μελών. Η προστασία των προσωπικών δεδομένων με τη σειρά της θα ενισχυθεί και αυτή. Νομίζω λοιπόν ότι η κατάληξη της προσπάθειας την οποία ξεκινήσαμε είναι θετική. Η νομική βάση της Europol έχει προσαρμοστεί στη συνθήκη της Λισαβόνας και οι στόχοι για τη μεταρρύθμιση της Europol έτσι ώστε να καταστεί πιο υπόλογη, αποτελεσματική και αποδοτική έχουν οι στόχοι αυτοί επιτευχθεί πλήρως. Θα ήθελα επίσης να σας παραπέμψω και στις δηλώσεις τις οποίες έκανε προς το Συμβούλιο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τις οποίες θα ήθελα να τονίσω και σήμερα. Η πρώτη άπτεται της διακυβέρνησης της Europol. Είμαστε πεπισμένοι μεν για τα πλεονεκτήματα της δημιουργίας ενός εκτελεστικού συμβουλίου για τη Europol και για άλλες εξωτερικές υπηρεσίες. Θα συνεχίσουμε να παρακολουθούμε την κατάσταση στις εξελίξεις γύρω από τη διακυβέρνηση της Europol και θα δούμε μετά από δύο χρόνια εάν απαιτούνται περαιτέρω προτάσεις. Η δεύτερη ανησυχία είναι η ανάγκη διασφάλισης συνοχής, συνεκτικότητας του πακέτου για τις αλλαγές στους κανόνες προστασίας δεδομένων και του κανονισμού λειτουργίας της Europol. Η επερχόμενη λοιπόν αυτή μεταρρύθμιση θα πρέπει να διασφαλίζει την συμβατότητα και να αποτρέπει τις επικαλύψεις του παρελθόντος θα πρέπει να είναι σαφές ότι ε, τα συμβούλια συνεργασίας στα πλαίσια αυτά, αυτής της ρυθμίσεως ε, θα μπορούν να ελέγχονται από το νέο σχετικά όργανο την υπηρεσία προστασίας δηλαδή προσωπικών δεδομένων. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ Επίτροπε. Δεν βλέπω την κυρία Χολμάγερ. Α, υπήρξε κάποια αλλαγή. Ποιος θα πάρει τη θέση της. Ο κύριος Βέρ θα πάρει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Η ασφάλεια των Ευρωπαίων πολιτών δοκιμάζεται και πάλι για διάφορους λόγους. Δεν επενδύσαμε πολύ στην άμυνα και ως εκ τούτου αντιμετωπίζουμε τώρα πολλές απειλές ε, για την ασφάλειά μας. Το βλέπουμε ε, στη Ρωσία, το βλέπουμε στον ε, ανταγωνισμό με την Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία είναι η μεγαλύτερη οικονομική δύναμη. Είναι πολύ σημαντικό σήμερα μετά από τριετής διαπραγματεύσεις να καταλήξουμε σε συμφωνία για την Europol. Χαίρομαι διότι σήμερα μπορούμε πλέον να ψηφίσουμε το νέο κανονισμό. Η Europol έτσι θα αποκτήσει περισσότερες αρμοδιότητες στην πάλι ενάντια στην τρομοκρατία. Η Europol θα μπορέσει επίσης να συστήσει ειδικέ μονάδες και η συνεργασία μεταξύ Europol και κρατών μελών θα βελτιωθεί πολύ. Είμαι περήφανος για την πολιτική μου ομάδα, η οποία τάχθηκε υπέρ της βελτιωμένης συνεργασίας με την Europol και φρόντισε γι' αυτό. Ενισχύσαμε την Europol και τώρα ε, έχουμε καλύτερο νομικό πλαίσιο. Οι πολίτες θα είναι περήφανοι για μας. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ για τους σοσιαλιστές Βάιντεν Τρία λεπτά. Αύριο είναι μεγάλη μέρα. Ε, σε δεύτερη ανάγνωση θα εγκρίνουμε τον κανονισμό για την Europol μετά από περισσότερο από τρία χρόνια και πάνω από 80 συνεδριάσεις. Ήταν επίπονη η διαδικασία και ο συνάδελφος Δίας Δεμέρα με μεγάλη συναδελφικότητα τα συντώνησε όλα αυτά ή και η συνάδελφος και θέλω να ευχαριστήσω και όλους τους κοιόδης που συνεργάστηκαν γιατί το εργασιακό κλίμα ήταν πολύ καλό. Σε ό,τι αφορά τις διατάξεις έχουν σύνδεση με τη συνθήκη της Λισαβόνας φροντίζοντας παράλληλα για την ασφάλεια των πολιτών ε, μειώνεται η γραφειοκρατία στη διασυνοριακή συνεργασία και έτσι θα είναι πιο αποτελεσματική πάλι κατά του οργανωμένου εγκλήματος και της τρομοκρατίας. Ο κανονισμός αυτός μπορεί να κάνει τις δομές της Europol πιο αποτελεσματικές και δημοκρατικές, ενισχύοντας τον κοινοβουλευτικό έλεγχο και ε, εισάγοντας και σημαντικές ε, διατάξεις για την προστασία των δεδομένων. Ο κοινοβουλευτικός έλεγχος μαζί με τα εθνικά κοινοβούλια είναι σημαντικό να ε, λαμβάνει η χώρα. Είναι σημαντική αυτή η νομική πράξη διότι εδώ είναι στο επίκεντρο η συνεργασία με τα εθνικά κοινοβούλια και τα ε, όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα θεσμικά όργανα και νομίζω ότι αυτό θα μπορέσει να αποτελέσει υπόδειγμα και για άλλες μορφές κοινοβουλευτικής συνεργασίας, γιατί εκεί το ευρωπαϊκό εγχείρημα έχει αδυναμίες. Σημαντικό είναι επίσης ότι καταφέραμε και στην τελευταία συνεδρίαση του Κοινοβουλίου για το πακέτο προστασίας δεδομένων. Ε, σημαντικό ήταν λοιπόν το γεγονός ότι μπορέσαμε να συνδέσουμε τις νεότερες εξελίξεις με την ανάγκη προστασίας δεδομένων. Θα ενισχυθεί και ως προς αυτό η Europol και θα εξασφαλιστεί αποτελεσματικότερη συνεργασία με αποδοχή των αρχών και θα υπάρχει μεγαλύτερη προθυμία για ανταλλαγή δεδομένων και διαβίβαση δεδομένων. Ε, σημαντικό είναι επίσης η σχέση πλέον Europol και SIPOL. Ε, εμείς πιστεύουμε ότι θα πρέπει να ενισχυθεί η εστίαση του κάθε οργανισμού. Αυτή τη ρεαλιστική προσέγγιση την ακολουθήσαμε και σε άλλους τομείς και στο παρατηρητήριο ε, που υπάρχει και που νομίζω θα έπρεπε να παίξει καλύτερο ρόλο, αλλά επίεζε ο χρόνος και έπρεπε να λάβουμε μια απόφαση. Ε, τελικά νομίζω ότι ο κανονισμός είναι καλός και βελτιώνεται η λειτουργία της Europol προς το συμφέρον των πολιτών. Δημιουργείται και μια βάση για περαιτέρω βήματα ολοκλήρωσης της αστυνομικής συνεργασίας που βεβαίως είναι τόσο απαραίτητη. Ο κύριος e παρακαλώ για δύο λεπτά. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε. Χρειάζεται η Europol να αντιμετωπίσει νέες προκλήσεις. Σήμερα μετά από μακριές διαπραγματεύσεις, επιτέλους έχουμε μια νέα εντολή για να αντιμετωπίσουμε τις τεράστιες ε, προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε. Υπό τον κύριο Wainwright, η Europol έχει γίνει ένας κόμβος που αντιμετωπίζει και παρέχει πληροφορίες σε όλη την επικράτεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εδώ θα δώσουμε τα νομικά εργαλεία στη Europol ε, έτσι ώστε να μπορεί να να αντιμετωπίσει με ταχύτητα αυτές τις προκλήσεις και να ακολουθήσει και τα εξαιρετικά υψηλά επίπεδα προστασίας προσωπικών δεδομένων που εμείς εδώ ε, συμφωνήσαμε. Θα πρέπει να υπάρχει λογοδοσία μέσω της ε, παρακολούθησης από τα Εθνικά Κοινοβούλια έτσι ώστε να είναι αξιόπιστες οι διοκτικές αρχές την Ευρωπαϊκή Ένωση. Επίσης έχουμε τη μονάδα την σχετική για το διαδίκτυο η οποία θα πρέπει να ενισχυθεί μια και οι εγκληματίες χρησιμοποιούν τα κοινωνικά δίκτυα για να προσελκύσουν. Το Twitter και οι λογαριασμοί του ε, είναι λογαριασμοί οι οποίοι θα πρέπει να παρακολουθούνται και όταν έχουμε περιεχόμενο τέτοιου είδους αμέσως να φροντίζουμε να κατεβαίνει. Γιατί πολύ συχνά οι πάροχοι υπηρεσιών ε, θεωρούν πως δεν έχουν την ευθύνη για το περιεχόμενο αυτό δεν είναι το FBI βέβαια η Europol, αλλά θα πρέπει να συνεχίσει να είναι αυτός ο κόμβος ε, ανταλλαγή πληροφοριών για όσους εργάζονται στις διοικητικές αρχές. Τρομοκρατία, ε, σοβαρό έγκλημα, πολύ συχνά είμαστε δύο βήματα πίσω από τους εχθρούς μας και ο κανονισμός αυτός θα κλείσει σε μεγάλο βαθμό αυτό το κενό. Η Europol έκανε την Ευρώπη και το Ηνωμένο Βασίλειο πιο ασφαλή για περίπου 20 χρόνια και ο κύριος Δίας Δεμέρα θα πρέπει και θα το πω, σας συγχαίρω για τον τρόπο με τον οποίο επιμείνατε έτσι ώστε το εργαλείο αυτό να βοηθήσει την Europol να συνεχίσει τη μάχη που δίνει κατά του εγκλήματος της τρομοκρατίας και όλων των ειδών τα λαθρεμπόρια όπως επίσης και της σεξουαλικής εκμετάλλευσης παιδιών. Ο κύριος Πίτερσον από τους Φιλελεύθερους παρακαλώ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Να ξεκινήσω ευχαριστώντας τον εισηγητή και τις υπηρεσίες ε, για την εξαιρετική τους πρόταση. Η διαδικασία αυτή ήταν μια μακρόχρονη διαδικασία και νομίζω ότι στο τέλος η Europol θα είναι πολύ καλύτερα εξοπλισμένη στην καταπολέμηση του σοβαρού εγκλήματος και της τρομοκρατίας. Θα ήθελα να ενισχυθεί ακόμα περισσότερο η Europol θα ήταν θετικό να είναι σε θέση η υπηρεσία αυτή να αποκτήσει περισσότερες αξουσίες και αρμοδιότητες στον τομέα της συλλογή πληροφοριών και γιατί όχι να υπάρχει ανταλλαγή πληροφοριών υποχρεωτική ανάμεσα στα κράτη-μέλη. Να μην μπορούν να συγκρατούν πληροφορίες στα κράτη-μέλη που θα μπορούσαν να φανούν χρήσιμες σε άλλες χώρες. Ο διαμεθοριακός χαρακτήρας των επιθέσεων των τρομοκρατικών στις Βρυξέλλες και στο Παρίσι αποδεικνύει ότι η συνεργασία των αστυνομικών δυνάμεων είναι καθοριστική για την καταπολέμηση της τρομοκρατικής απειλής. Δυστυχώς μέχρι τώρα δεν τα έχουμε καταφέρει. Οι τρομοκράτες ε, του Νοεμβρίου στο Παρίσι είχαν έρθει στις Βρυξέλλες, τους είχαν σταματήσει στα σύνορα αλλά τους άφησαν μετά γιατί η γαλλική αστυνομία πάρα πολύ απλά δεν είχε τις φωτογραφικές πληροφορίες έτσι ώστε να τους συλλάβει. Πρέπει λοιπόν να υπάρξει καλύτερη ανταλλαγή πληροφοριών ανάμεσα στα κράτη-μέλη. Είναι η βασική προϋπόθεση έτσι ώστε να αποφύγουμε μελλοντικού τύπου επιθε... μελλοντικές επιθέσεις τέτοιου τύπου. Θα πρέπει να δράσουμε πριν υπάρξουν νέες επιθέσεις και για να το πετύχουμε η προσπάθεια πρέπει να είναι κοινή. στο δημοψήφισμα οι Δανείοι είχαν ψηφίσει την αποχώρησή τους από τη Europol γιατί δεν ήταν ικανοποιημένοι από τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούσε. Αλλά ελπίζω με τη νέα ρύθμιση η Δανία να επανέλθει και υπάρχουν και οι διμερείς και παράλληλες βέβαια συμφωνίες οι οποίες όμως δεν είναι καλή λύση. Εύχομαι λοιπόν ό,τι καλύτερο για τη νέα προσπάθεια ενίσχυσης της Europol. Ευχαριστώ πολύ από την ΚΟΕ κυρία Ένστ για 1,5 λεπτό. Ευχαριστώ. Να ευχαριστήσω καταρχήν τον εισηγητή ο οποίος ε, συνεργάστηκε επικοδομητικότατα παρά τις διαφορετικές θέσεις. Το αποφασιστικό για μας ήταν τι θέλαμε από την αστυνομία. Αυτό είναι το κύριο ερώτημα. Ε, με την Europol χρειάζεται να υπάρχει συντονισμός και θέλουμε οι πολίτες να προστατεύονται αποτελεσματικά στα θεμελιώδη δικαιώματά τους, να αντιμετωπίζεται αποτελεσματικά το έγκλημα και να ε, υπάρχει συνεργασία υπό δημοκρατικό έλεγχο. Αυτό ήταν το βασικό. Ε, υπάρχουν ε, δυνατότητες για βελτίωση ε, και συνολικά δεν είμαστε ικανοποιημένοι. Ε, όταν, για, να έχουμε αποτελεσματική διασυνοριακή συνεργασία θα πρέπει τα αδικήματα ε, στον κατάλογο να ε, διευρυνθούν, να διευρυνθεί ο κατάλογος των αδικημάτων. Δηλαδή, επίσης με το Internet Referral Unit δημιουργείται ένα όργανο στην πράξη χωρίς νομική βάση και στήριξη με το οποίο σε τελευταία ανάλυση ε, μπορεί να λαμβάνονται αυθαίρετες αποφάσεις για τις πληροφορίες από το ίντερνετ. Και υπάρχει και συνεργασία με ιδιωτικούς φορείς ε, που θα αποφασίσουν τι ε, είναι σημαντικό και τι δεν είναι στη διαβίβαση των δεδομένων. Επίσης ε, υπάρχει θέμα με τον κοινοβουλευτικό ε, έλεγχο. Περιμέναμε περισσότερα εδώ. Δεν υπάρχει επαρκής κατοχυρωσή της. Υπάρχουν ε, ε, πολλά, πολλές ελλείψεις και γι' αυτό συνολικά ψηφίζουμε κατά. Ευχαριστώ πολύ ο κύριος Τυρίκα Ώρας από τους Πράσινους. Σας ευχαριστώ πολύ. Η Europol είναι η ευρωπαϊκή υπηρεσία που στηρίζει τις εθνικές διοκτικές αρχές στη μάχη κατά του διεθνούς εγκλήματος και της τρομοκρατίας. Οι πιο πρόσφατες τρομοκρατικές επιθέσεις έχουν αυξήσει την ανάγκη που υπάρχει να δημιουργηθεί μια πιο ισχυρή Ευρωπαϊκή Αστυνομική Αρχή με μεγαλύτερες δυνατότητες για μεθοριακή συνεργασία και ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ κρατών μελών. Στα πλαίσια αυτά ήταν απαραίτητο να πρικοδοτήσουμε την Europol με τα μέσα για να στηρίξει τα κράτη-μέλη στην πρόληψη, στην ανάλυση και στην έρευνα που γίνεται για εγκλήματα σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Όμως, όσο πιο δυνατή είναι η Europol, τόσο περισσότερο θα πρέπει να είναι και ο κυβερνητικός, με συγχωρείτε, ο κοινοβουλευτικός έλεγχος της δράσης της. Και θα πρέπει να έχουμε και περισσότερα νομικά εχέγγυα, έτσι ώστε να μην υπάρχει μία ε, παρακολούθηση ανεφλόγου μαζική των ε, ε, συμπολιτών μας και μια χωρίς λόγο συλλογή προσωπικών δεδομένων που θα παραβιάζει τα θεμελιώδη δικαιώματα όσων εμείς υπηρετούμε. Η Europol δραστηριοποιείται μέσα στα σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το οργανωμένο έγκλημα δεν σταματά στα σύνορά μας και γι' αυτό είναι απαραίτητο να έχουμε καλύτερη συνεργασία με τρίτες χώρες όπως επίσης και με οργανώσεις διεθνείς του χώρου. Ο κανονισμός που συζητάμε έχει στόχο να ενισχύσει τη Europol και να αποφύγουμε κάποιους κινδύνους που έχουμε, να έχουμε αυξημένη αστυνομική παρουσία και αστυνόμευση της πρωτοπικής μας ζωής. Και υπάρχουν κάποια θέματα που ανησυχούν την ομάδα μου, για παράδειγμα το γεγονός πως εκτελεστικός διευθυντής της Europol δεν λογοδοτεί άμεσα στο ε, Ευρωπαϊκού Κοινοβούλιο αλλά στο δικό του Συμβούλιο. Και επίσης η νομική βάση ε, για τη μονάδα, το Internet Referral Units, ε, ε, αλλάζει από αυτό που είχαμε από 1η Ιουλίου του 2015 και γι' αυτό διατηρείται η τροπολογία μας για να διατηρηθεί όπως είχε συμφωνηθεί και να μην αποτελεί κομμάτι ε, διαφορετικής νομικής, ε, νομοθετικής πρότασης, αλλά να παραμείνει στο κείμενο που είχαμε εγκρίνει τότε. Τώρα, ευχαριστώ τον συνάδελφο, ο οποίος έκανε ε, προσπάθειες να βελτιώσει το κείμενο. Εμείς θα υπερψηφίσουμε την τροπολογία που υποβάλλουμε, αλλά θα στηρίξουμε και το κείμενο του κυρίου Διασμέρα στο σύνολό του, γιατί είναι απαραίτητο και δεν υπάρχει εναλλακτική λύση. Θέλουμε καλύτερη και μεγαλύτερη και ενισχυμένη συνεργασία μεταξύ των ευρωπαϊκών διοκτικών αρχών έτσι ώστε να υπάρχει συμμόρφωση με τον νόμο και να έχουμε καλύτερη ανταλλαγή πληροφοριών με τρίτες χώρες στις ε, προσπάθειες που γίνονται να καταπολεμήσουμε το οργανωμένο διεθνές έγκλημα. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Μαχ, επόμενο για 1,5 λεπτό. Κυρίες και κύριοι, όταν ψηφίσουμε την πρόταση αυτή, Μία πρόταση θα έχουμε να ψηφίσουμε. Τη, την πρότασή μου για απόρριψη αυτής ε, της διάταξης, ε, η οποία υπευλήθη εξ ονόματος της ομάδας μου, διότι δεν είχαμε τη δυνατότητα να ε, υποβάλουμε τροπολογίες για το κείμενο. Αυτό σημαίνει άρνηση της κοινοβουλευτικής δημοκρατίας. Πρόσφατα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπέβαλε διαφορετικό σχέδιο και το βασικό ήταν η συνένωση Europol και Σύπολ. Αυτό ε, είναι εκτός συζήτησης στο Κοινοβούλιο. Ε, άλλαξε τελείως η Europol και έγινε νέος οργανισμός. Ε, δημιουργήθηκε δηλαδή ε, ένας αστυνομικός οργανισμός, ε, μια μυστική τροποντινά αστυνομία για την Κομισιόν και το Συμβούλιο. Ε, η Κομισιόν θα μπορεί έτσι να διαβιβάζει δεδομένα τα οποία συλλέγει η Europol προς άλλους ε, οργανισμούς. Ε, συμφωνήσατε ιδιωτικές εταιρείες και αεροπορικές εταιρείες αυτομάτως να μπορούν να διαβιβάζουν δεδομένα, αριθμούς λογαριασμών, διευθύνσεις, ονόματα προσώπων και αυτή η νέα Europol θα μπορεί επίσης να διαβιβάζει σε ιδιώτες τα ε, δεδομένα αυτά. Θα βρίσκεται δηλαδή εκτός δικού μας ελέγχου. Το σχέδιο ε, προσχηματικά αναφέρεται σε κάποιο μορφής έλεγχο, αλλά ε, νομίζω ότι αυτό που ζητείτε ε, είναι πολύ περιορισμένο ισότητα ανδρών και γυναικών ενώ πίσω κρύβεται ένα θεσμικό όργανο πάρα πολύ επικίνδυνο. Καταψηφίστε παρακαλώ. Ευχαριστώ. Ο κύριος ε, Πρέτσελ για ένα λεπτό παρακαλώ. Ο προηγούμενος ομιλητής ξεπέρασε το χρόνο ομιλίας. Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, όλοι, ή τουλάχιστον η πλειοψηφία στο κοινοβούλιο αυτό, Εορτάζεται σήμερα ένα μεγάλο πλήγμα κατά της τρομοκρατίας στην Ευρώπη, ε, εφοδιάζοντας με νέες αρμοδιότητες ε, την Europol. Ανταλλαγή δεδομένων ε, διευρύνεται έτσι. Υπάρχει η υποστήριξη των σκιωδών αλλά ίσως αυτό πρέπει να μας ε, κάνει να ανησυχήσουμε διότι μπορεί να υπάρχει υπερβολική συνένεση υπέρ της υπερβολικής διαβίβασης δεδομένων. Οι εκπρόσωποι της λεγόμενης ε, φιλελεύθερης ομάδας δηλώνει ότι δεν υπάρχει αρκετή ε, υποχρέωση διαβίβασης δεδομένων και ότι θα πρέπει αυτή να διευρυνθεί ακόμη περισσότερο. Αυτά είναι αστεία πράγματα. Δεν είμαστε σε θέση στην Ευρώπη τους κανόνες που είχαμε θέσει στο παρελθόν δηλαδή προστασία εξωτερικών ε, συνόρων, ε, Σέγγεν, ε, Συμφωνία του Δουβλίνου. Αυτούς τους κανόνες που έχουμε θεσπίσει δεν μπορούμε να τους εφαρμόσουμε στο έδαφος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και τώρα θέλετε να δημιουργήσετε και νέους κανόνες για να καταπολεμήσετε προβλήματα που δημιουργήθηκαν. Γιατί, γιατί απλούστατα δεν μπορέσαμε να εφαρμόσουμε τους παλιούς κανόνες. Δεν μπορεί να είναι σοβαρά αυτή η πρόθεση του Κοινοβουλίου. Θα πρέπει κάποια στιγμή να ανατρέξουμε στους παλιούς κανόνες, να ανταποκριθούμε σε αυτούς, να τους εφαρμόσουμε και όχι να θεσπίζουμε συνεχώς καινούριου επειδή προβλήματα που προκύπτουν επειδή δεν ε, αντιμετωπίσαν τους παλιούς. Ο κύριος Αργιανόπουλος, παρακαλώ, ένα λεπτό. Η Ευρωπόλ επανειδρύεται σαν ευρωενωσιακό όργανο ενισχύοντας και διευρύνοντας το έπακρο τον κατασταλτικό της ρόλο επεμβαίνει στα κράτη μέλη με την ίδρυση εθνικών κέντρων διασύνδεσης με την Ευρωπόλ. έχει το δικαίωμα να απαιτεί από αυτά την κίνηση ποινικών διώξεων σε ευρύτατη γκάμα αδικημάτων. με το βολικό πρόσχημα κατά καταπολέμησης τρομοκρατίας γίνεται κέντρο φακελώματος τεράστιας έκτασης προσωπικών δεδομένων μέχρι και για τις κοινωνικές συναναστροφές του καθενός. κόμβος ανταλλαγής αυτών των πληροφοριών με αρχές ασφαλείας και μυστικές υπηρεσίες των κρατών μελών και τρίτων χωρών ιδίως των ΗΠΑ ακόμα και με ιδιώτες όπως παραδείγματος χάρη με την παρακολούθηση του διαδικτύου σε διασύνδεση με τους επιχειρηματικούς ομίλους του κλάδου. οι ισχυρισμοί σας για δίθεν προστασία των δεδομένων και κοινοβουλευτική λογοδοσία αποτελούν κοροϊδία και άλοθη νομοποίηση τη κατασταλτικής αυτής δράσης. στο επίκεντρο του φακελώματος βρίσκεται η πολιτική και κοινωνική δράση με στόχο την αντιμετώπιση των λαϊκών κινημάτων ενάντια στην αντιλαϊκή πολιτική ευρωπαϊκής ένωσης και κυβερνήσεων. το εργατικό λαϊκό κίνημα μπορεί ενισχύοντας την πάλη του να αντιμετωπίσει και τους κατασταλτικούς μηχανισμούς θωράκισης εξουσίας των μονοπωλίων την οποία πρέπει να ανατρέψει. Ζητείτε μία μπλε κάρτα. Μπορείτε να απαντήσετε, επιθυμείτε να απαντήσετε. Est-ce que vous acceptez Pane kolego, já nevím, jestli jste to nařízení nebo tento dokument vůbec četl. Ε, δεν ξέρω αν διαβάσατε τον κανονισμό, αν γνωρίζετε το κείμενο. Γι' αυτό με ενδιαφέρει η απάντησή σας. Μπορείτε να μου πείτε και να μου εξηγήσετε Πώς γίνεται κατασταλτικός οργανισμός η Europol. Έχετε πάει να επισκεφθείτε την Europol. Ξέρετε πώς λειτουργεί. Παρακαλώ απαντήστε με. Ευχαριστώ. Δεν είναι ανάγκη κάποιο να επισκεφθεί τα γραφεία της Europol για να καταλάβει το χαρακτήρα της. Το ίδιο ακριβώς το κείμενο είναι αυτό το οποίο δίνει αυτόν τον κατασταλτικό χαρακτήρα. Διευρύνεται το αντικείμενο των πληροφοριών τις οποίες συλλέγει σε μια τεράστια γκάμα αν το διαβάσει κανένας προσεκτικά για όλες τις προσωπικές συνήθειες δραστηριότητες του κάθε ανθρώπου. αυτό βεβαίως αν κάποιος επίσης το διαβάσει προσωπικά θα καταλάβει ότι ιδιαίτερα επικεντρώνεται στην κοινωνική πολιτική και συνδικαλιστική δραστηριότητα γιατί ακριβώς εκεί βρίσκεται ο φόβος αυτών που θέλουν να ελέγξουν αυτή την κοινωνική δραστηριότητα. Αυτό είναι ο κατασταλτικός χαρακτήρας της europol. Η κυρία... Κύριε Πίτροπε, κυρία Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, εκπλήσωμε με ορισμένες αντιδράσεις ε, συναδέλφων και από το κέντρο και από αριστερά ε, που δείχνουν άγνοια. Εδώ έχουμε μια συνεργασία και συντονισμό των διαφορετικών ε, αστυνομιών και ε, υπηρεσιών ασφαλείας. Στο Internet ε, Referral Unit δεν ε, γίνονται αυθαιρεσίες. Αντίθετα απομακρύνονται αποτρόπαια εγκλήματα από το διαδίκτυο για να μην οδηγούν σε ε, ε, κακοποίηση παιδιών ε, και άλλα εγκλήματα, ούτε να τα βλέπουν παιδιά. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό και όταν υπάρχουν αμφιβολίες μπορεί κανείς να προσφύγει στα δικαστήρια. Αυτό σημαίνει κράτος δικαίου. Επίσης μπορεί κανείς να πει ότι η Europol δεν έχει δικαίωμα ε, να επιβάλλει μέτρα απέναντι σε έναν οργανισμό. Αυτό θα πρέπει να το κάνουν οι ε, αρμόδιοι ε, εθνικοί φορείς ε, δεν ξέρω, νομίζω ότι πολλοί συνάδελφοι δείχνουν άγνοια. Εις ό,τι αφορά την αυθαιρεσία ε, στη διαβίβαση των δεδομένων, όχι. Ε, όλα αυτά είναι κρυπτογραφημένα. Υπάρχουν πάρα πολλοί συγκεκριμένοι περιορισμοί για, στη διαβίβαση των δεδομένων. Νομίζω ότι η μεταρρύθμιση της Europol έγινε επιτυχώς. Θέλω να συγχαρώ τον εισηγητή Αγκουστίν Διαστεμέρα και τους Σκιώδης. Ε, ε, νομίζω και ε, ο συνάδελφος από την Άλντε έχει δίκιο που λέει ότι χρειαζόμαστε περισσότερη ανταλλαγή δεδομένων γιατί το έγκλημα δεν γνωρίζει σύνορα και βεβαίως συγχαίρω και για την πρόταση της Κομισιόν. Θα ήθελα η Κομισιόν να διαθέσει και περισσότερο προσωπικό για, στη Europol, γιατί ο αριθμός 30 δεν επαρκεί. Ελπίζω όμως, νομίζω όμως ότι γενικά υπήρξε επιτυχία και ε, αυτό που είπατε για τις τροπολογίες, βεβαίως υπήρξαν και κατατέθηκαν πάρα πολλές τροπολογίες. Δυστυχώς εσείς συνάδελφοι δεν, δεν συμμετείχατε. Η κυρία Γκόμες για δύο λεπτά. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα καταρχήν να χαιρετήσω τις προσπάθειες που έκανε και ο κύριος Δίας Δεμέρα και οι υπόλοιποι εισηγητές εδώ και πάνω από δύο χρόνια διαπραγματεύσεων για τα κράτη-μέλη δεν επιθυμούσαν να εισάγουν αυτή την αστυνομική συνεργασία στην αρχή στα κείμενά μας. Είναι πολύ σημαντικό το ότι αλλάζει αυτή η νοοτροπία, αλλάζουν οι πρακτικές που ακολουθούμε και μετά τις τρομοκρατικές επιθέσεις που είχαμε στις Βρυξέλλες και στο Παρίσι ε, πρέπει να σας πω πως αντιμετωπίσαμε το βασικό πρόβλημα της έλλειψης συνεργασίας μεταξύ αστυνομικών αρχών και μεταξύ κρατών μελών και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, κάτι το οποίο ευνοεί το οργανωμένο έγκλημα που είναι όλο και περισσότερο διεθνές. Ο κανονισμός αυτός ε, δημιουργεί τον δημοκρατικό έλεγχο από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και από τα Εθνικά Κοινοβούλια. Και θα πρέπει να απαιτήσουμε εμείς από τις κυβερνήσεις μας ε, να συνεργαστούν με την Europol και να ανταλλάσσουν πληροφορίες και βέβαια θα πρέπει να προστατεύσουμε τους πολίτες μας. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κατάφερε να επιβάλλει ε, το σεβασμό για τις αρχές της προστασίας των προσωπικών δεδομένων. Αυτό είναι το πιο ουσιαστικό και νομίζω ότι θα πρέπει η διαλειτουργικότητα των βάσεων δεδομένων επίσης να εξασφαλιστεί και για το IRU. Αναγνωρίζετε εδώ πως η Europol είναι ένα εργαλείο απαραίτητο στη μάχη κατά της τρομοκρατίας του οργανωμένου εγκλήματος. Το είδαμε αυτό στο τι συνέβη με ε, την ρωσική μαφία και το δίκτυό της στην Πορτογαλία που καταφέραμε ε, να διαλύσουμε παρόλη την παρουσία που είχαν στις ποδοσφαιρικές ομάδες στη χώρα μου. Και πρέπει να σας πω πως τα κράτη-μέλη εξακολουθούν να φέρουν την ευθύνη σε τοπικό επίπεδο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο στη μάχη κατά της ε, τρομοκρατίας και του οργανωμένου εγκλήματος και χρειάζεται να υπάρχει συνεργασία μεταξύ των διαφόρων υπηρεσιών, όπως επίσης και μια διασύνδεση ε, των αποκρίσεων που δίνουμε σε εσωτερικό και εξωτερικό επίπεδο. Θα πρέπει τα κράτη-μέλη να συνεχίσουν να εργάζονται μέσω συγκεκριμένων προγραμμάτων και όπως είδαμε και με το θέμα των φορολογικών παραδείσων να συνεχίσει η μεταξύ μας συνεργασία. Θα πρέπει λοιπόν να δούμε πώς μπορούν όλα αυτά να εφαρμοστούν γιατί συνέχεια θα αποκαλύπτουμε όλο και περισσότερο δίκτυα εγκληματικά με ε, τρομοκρατικές επίσης διαστάσεις. Ευχαριστώ πολύ. Στίβενς για ένα λεπτό. Αγαπητοί συνάδελφοι, η αντιπροσωπεία μου είναι ικανοποιημένη από την ε, κατάληξη των διαπραγματεύσεων. Η Ευρωπόλ θα μπορέσει να συνεργαστεί στενότερα με τις υπόλοιπες δυνάμεις και έτσι θα είναι καλύτερα προετοιμασμένη αν χρειαστεί να βοηθήσει τις χώρες να καταπολεμήσουν το οργανωμένο έγκλημα και την τρομοκρατία. θα μπορούσαμε σαν παράδειγμα να ειδοποιήσουμε για την κυκλοφορία ύποπτων tweet ε, ιδιαίτερα σε σχέση με τους τζιχαντιστές υπάρχει δυνατότητα να λειτουργήσει η Europol καλύτερα και να είναι πιο ενημερωμένη. θα έχει επίσης ε, ένα σύστημα διαχείρισης δεδομένων το οποίο θα είναι πολύ πιο σύγχρονο και πολύ πιο ικανό σύμφωνα πάντα ε, με ε, τα βέλτιστα τεχνικά χαρακτηριστικά που απαιτούνται. Είναι ένα πολύ θετικό βήμα. Ο κύριος Ντεπρέ έχει το λόγο. Πρόεδρε, Επίτροπε, Είμαι πεπισμένος ότι είναι θετική η πρόταση που μας υποβάλλεται σήμερα μετά από χρόνια δουλειάς. Υπάρχουν ξεκάθαροι κανόνες που θα ενισχύσουν το κέντρο καταπολέμησης της τρομοκρατίας, βελτιώνοντας την ανταλλαγή ε, ενημερωτικών στοιχείων. Υπογραμμίζεται ότι θα μπορεί και να ανταλλάσσει πληροφορίες η Europol με ιδιωτικές επιχειρήσεις, κάτι το οποίο θα μπορεί, θα επιτρέπει σαν παράδειγμα στη Europol να ζητεί από την Google ή από το Facebook να διαγράφει σελίδες οι οποίες υμνούν ε, το Ισλαμικό κράτος. Θα πρέπει φυσικά να είναι ενημερωμένη η κοινοβουλευτική κάθε χώρας. Καταρχάς πρέπει όμως να πω στο αρνητικό επίπεδο ότι σε σχέση με την εκκίνηση των ποινικών διαδικασιών δεν έχει τη δυνατότητα πρωτοβουλίας και δεν υπάρχει έστω και σε εμβριακή κατάσταση μία πρόταση για τη δημιουργία μιας Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Συλλογής Πληροφοριών. Θα μετανιώσει το Συμβούλιο στο μέλλον γι' αυτό. Άντερσον. όλες οι αρχές θα πρέπει να υφίστανται ε, τον αδημοκρατικό έλεγχο, τον κοινοβουλευτικό έλεγχο. Εμείς στο ΣΥΝΦΕΙΝ κατανοούμε την ανάγκη συνεργασίας ε, ανάμεσα στις διάφορες χώρες, ιδιαίτερα στον τομέα της τρομοκρατίας, της λαθρεμπορίας ναρκωτικών και του τράφικινγκ αλλά η απομάκρυνση της μικτής επιτροπής ελέγχου ε, που είχε την δυνατότητα να βλέπει τον τρόπο με τον οποίο ε, λειτουργούσε η ε, Europol δεν θα μπορεί να λειτουργεί στο μέλλον με τον ίδιο τρόπο. Ιδιαίτερα γιατί η πρόταση αυτή θα δώσει τη δυνατότητα στη Europol να, να διαχειρίζεται πάρα πολύ ε, μεγάλες ποσότητες προσωπικών δεδομένων. Όταν κάποιος αναλαμβάνει περισσότερες ευθύνες πρέπει να έχει ε, και περισσότερες ευθύνες ο ίδιος για τη διαχείρισή τους. Ο κύριος Άλμπρεχτ, δύο λεπτά. Αξιότιμη κυρία Πρόεδρε, αξιότιμη κυρία Επίτροπε, θέλω να ευχαριστήσω τον εισηγητή, κύριο Ντίας Δεμέρα, για την καλή δουλειά Ήδη αναφέρθηκε και από τους Σκιώδης ότι σημειώθηκαν μεγάλες πρόοδοι στον κανονισμό για την Europol και όλοι πρέπει να διαπιστώσουμε ότι πρόκειται για πρόοδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχουμε ένα νέο κανονισμό για την Europol που φροντίζει για περισσότερη Ευρώπη στον τομέα της δίωξης, αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Σημαντικό είναι επίσης ότι προβλέπονται σαφείς διατάξεις προστασίας δεδομένων που ε, θέλουμε να συνάδουν, συνάδουν με το πακέτο για την προστασία δεδομένων. Ε, αυτό δημιουργεί ασφάλεια στους πολίτες και δημιουργεί τη βάση νομιμοποίησης για τη λειτουργία καλύτερου συστήματος ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ αστυνομικών και δικαστικών ε, αρχών, διοκτικών εν προκειμένου και της Europol. Εγώ θα ήθελα, οι πράσινοι θα επιθυμούσαν αν σε δύο σημεία θα μπορούσαμε να είχαμε κάνει περισσότερα βήματα. Το ένα είναι κάτι που πρέπει να γίνει, πρόκειται για την, ε, την καλύτερη σύνθεση των ε, ομάδων έρευνας στη Europol, γιατί δεν μπορούμε να ε, στηριζόμεθα στα δεδομένα και στους κομπιούτερ αν θέλετε, αλλά οι υπάλληλοι επιτόπου θα πρέπει να έχουν καλύτερη δικτύωση ε, θα πρέπει δηλαδή να έχουν τα απαραίτητα μέσα πόρους οικονομικούς και ανθρώπινους για να δρουν αποτελεσματικότερα διασυνοριακά. Αυτό θα πρέπει να γίνει. Επίσης, σε ό,τι αφορά τη διαβίβαση πληροφοριών σε τρίτους ιδιώτες, θα έπρεπε να δημιουργηθεί ένα πλαίσιο ε, ε, δημοσίου δικαίου. Αυτό δεν γίνονται. Δηλαδή δεν αντιμετωπίζονται οι ιδιώτες όπως και οι κρατικοί φορείς. Εδώ είχαμε υποβάλει μια σχετική τροπολογία και αντίθετα με τους ε, δεξιούς συναδέλφους μας εμείς συμμετέχουμε στη διαδικασία και θέλουμε το κείμενο να βελτιωθεί. Κατά τα άλλα, νομίζω ότι είναι καλή η πρόταση για την Europol. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Φωνστόρχ. μισή λεπτό. Συζητούμε για μεταρρύθμιση της Europol. Η Europol θα συλλέγει δεδομένα και θα συνεργάζεται και θα τα ανταλλάσσει με δημόσιες και ιδιωτικές αρχές. Θα υπάρξει και μια, ένα, ένα ε, τμήμα έρευνας ε, το οποίο ε, θα μπορεί να έχει πρόσβαση σε ιδιωτικές και δημόσιες βάσεις δεδομένων, θα τις αποθηκεύει, θα τις συλλέγει, θα τις διαβιβάζει. Πρόκειται για πληροφορίες που αφορούν ένα σωρό δεδομένα από διπλώματα οδήγησης, διευθύνσεις, αριθμούς λογαριασμών, φωτογραφίες, ε, προηγούμενους ε, εργοδότες, ε, ε, ομόλογα, ε, σύνδεση με επιχειρήσεις, φορολογικά δεδομένα κλπ. Επίσης υπάρχει ενδιαφέρον σε σχέση με τον τρόπο ζωής του κάθε προσώπου, ενδεχόμενη χρήση ουσιών κλπ. Όλα αυτά λοιπόν συλλέγονται. Θα τα ξέρει όλα δηλαδή η Europol. Ε, στο όνομα της καταπολέμησης της τρομοκρατίας ε, ένα πράγμα μπορεί να, διατέξει, να διατρέξει κίνδυνο. Η ασφάλεια των δεδομένων όλων των πολιτών. Ευχαριστώ. Ο κύριος Επιτίδιος, ένα λεπτό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Μία από τις παρενέργειες της παγκοσμιοποίησεως είναι και η αύξηση των απειλών καταδοχών της Ευρώπης και η ποιοτική τους αναβάθμιση. Ε, οι απειλές αυτές είναι κυρίως η τρομοκρατία, η επιθέσει στον κυβερνοχώρο και το οργανωμένο έγκλημα. οι λαοί τη Ευρώπη αισθάνονται ανασφάλεια και υπονομεύεται η ασφάλεια των προσωπικών του δεδομένων. η ευρωπαϊκή αστυνομική υπηρεσία η europol είναι ο φορέας εκείνο ο οποίο καλείται να αντιμετωπίσει αυτέ τι απειλέ σε συνεργασία με τι αστυνομικέ και τι δικαστικέ αρχέ ε, των άλλων χωρών. για να μπορέσει να εκτελέσει με επιτυχία αυτή την αποστολή πρέπει να ανταλλάσσει πληροφορίε με αυτέ τις υπηρεσίε και με υπηρεσίε τρίτων χωρών και στο σημείο αυτό πρέπει να προσέξουμε ιδιαίτερα. Ε, ε, ε, επειδή αυτές οι πληροφορίες άπτονται και προσωπικών δεδομένων πρέπει πάση θυσία να εξασφαλιστεί ότι η απέτηση για την ασφάλεια δεν θα παραβιάζει τα ανθρώπινα δικαιώματα. πρέπει να παρέχονται πληροφορίες μόνο όταν είναι σχεδόν βέβαιο ότι ένας πολίτης είναι ύποπτος να εκτελέσει τρομοκρατικές ή άλλης φύσεως ενέργειες. και τέλος πρέπει να εξασφαλιστεί ότι οι πληροφορίες αυτές δεν θα χρησιμοποιηθούν για δίωξη πολιτικών αντιπάλων είτε από αντιδημοκρατικέ κυβερνήσει είτε από κυβερνήσει που έχουν αντιδημοκρατική ε, και καθεστωτική νοοτροπία. Ευχαριστώ. Ε, what are the crucial elements to our... Ποια είναι τα βασικά στοιχεία τα οποία πρέπει να χρησιμοποιήσουμε για να καταπολεμήσουμε τις τρομοκρατικές απειλές. Πολλοί από εμά υπογράμμισαν ότι η στενότερη συνεργασία είναι κάτι το θεμελιώδες και αυτό σημαίνει και καλύτερη και σωστότερη διαχείριση στη Europol. Η πρόταση είναι σωστή λοιπόν, θα μας δώσει τα προληπτικά μέτρα τα οποία απαιτούνται γιατί η πρόληψη είναι πλέον το κλειδί. Η Europol θα έχει καλύτερη πρόσβαση στα σχετικά στοιχεία τα οποία θα μπορεί να επεξεργαστεί πιο αποτελεσματικά και τα δεδομένα από τα κράτη-μέλη αλλά και από μη δημόσιες υπηρεσίες που και αυτά είναι χρήσιμα για την πρόληψη και την έρευνα. Το Internet Referral Unit θα παίξει ένα σημαντικό ρόλο στην καταπολέμηση της προπαγάνδας ε, και της ριζοσπαστικοποίηση online. Νομίζω ότι η συνεργασία με τους παροχείς ε, ίντερνετ θα ε, διώξει από το διαδίκτυο κάθε μορφή βίαιου περιεχομένου. Νομίζω ότι πρέπει να ενισχύσουμε τους κανόνες προστασίας όμως και των προσωπικών δεδομένων για να υπάρξει σωστή ισορροπία. Ενισχύσαμε τις δυνατότητες συνεργασίας της Europol και με άλλες ευρωπαϊκές υπηρεσίες για καλύτερες συνέργειες και αποτελεσματικότητα. Αυτό το οποίο ισχύει είναι ότι τα κράτη-μέλη πρέπει να μοιράζονται τις πληροφορίες με τη Europol Τότε μόνο θα δουλέψει το σύστημα, αλλιώς η Europol δεν θα μπορέσει να εκμεταλλευτεί όλες τις δυνατότητες. Θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Διάς Ντεμέρα για την αποφασιστικότητά του μέχρι τώρα. Η κυρία Κάουφμα, δυόμιση λεπτά. Σήμερα δίνουμε πράσινο φως στη μεταρρύθμιση της Europol και υπάρχουν πολύ σημαντικοί λόγοι γι' αυτό. Η εγκληματικότητα δεν γνωρίζει σύνορα, γι' αυτό υπάρχει ανάγκη ενίσχυσης ε, της Europol και της συνεργασίας με τις εθνικές αρχές και άλλους ε, οργανισμούς. Θα βελτιωθεί η ανταλλαγή δεδομένων και θα υπάρξουν σύγχρονες διοικητικές δομές. Στο μέλλον η Europol θα μπορεί να ε, ανταποκρίνεται καλύτερα στις απειλές και μέσω της σύστασης ειδικών μονάδων. Είναι σημαντικό για τη μεταρρύθμιση να έχουμε υψηλά ε, στάνταρ για τη διαβίβαση δεδομένων και τη δίωξη. Και αυτά τα στάνταρ θα ισχύουν για τη Europol. Ε, φωνές ε, μίσους ε, ε, στο ίντερνετ μπορεί να κάνουν μεγάλη ζημιά. Γι' αυτό θα πρέπει να εξαφανίζονται από το ίντερνετ το ταχύτερο δυνατόν. Ε, επίσης, το Internet Referral Unit τώρα αποτελεί, στηρίζεται σε στέρεη βάση. μπορεί να διασφαλίζεται η ανταλλαγή δεδομένων. Η βάση ε, για την αστυνομική συνεργασία ε, είχε ήδη ε, συσταθεί και είναι σημαντικό η μεταρρύθμιση της Europol να λειτουργεί βάσει των διατάξεων της συνθήκης της Λισαβόνας. Νομίζω ότι πρέπει να τονίσουμε ότι για πρώτη φορά σε οργανισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα υπάρξει δημοκρατικός έλεγχος ε, από ε, βουλευτές της Αρμόδιας Επιτροπής και από εκπροσώπους των Εθνικών Κοινοβουλίων. Όλα αυτά ε, δείχνουν ότι ο δημοκρατικός έλεγχος και η προστασία των δεδομένων δεν είναι σε αντίθεση αλλά πρέπει να συνάδουν το ένα με το άλλο. Ευχαριστώ πολύ τον κύριο Ευχαριστώ πολύ. Πρέπει να σας πω πως ο κανονισμός αυτός ε, θα αυξήσει την ασφάλεια για τους Ευρωπαίους πολίτες και για την Ευρώπη ολόκληρη. Είναι κρίμα που το κείμενο είναι τόσο ελαφρύ, γιατί αν δεν είχαμε και τα δραματικά γεγονότα πρόσφατα, ακόμα δεν θα είχαμε κλείσει τον κανονισμό όσοι είναι αντίθετοι με τον κανονισμό αυτό, με λανθασμένο τρόπο περιγράφουν τα όσα προσπαθεί να πετύχει ε, ως μια προσπάθεια κεντρική ε, καταπάτησης των προσωπικών ελευθεριών, ως ένα παράλογο βήμα ε, για να περιορίσουμε τις προσωπικές ελευθερίες. Όμως αυτή η υπηρεσία θα παρακολουθεί και το ίντερνετ με τον απαραίτητο δημοκρατικό έλεγχο που χρειάζεται. Και ούτε η άκρα αριστερά ούτε η άκρα δεξιά υπηρετούν τα συμφέροντα του κοινού υποστηρίζοντας το αντίθετο. Η κυρία Βίξτρομ, ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Πιστεύω πως εδώ έχουμε κάτι καλό και επιτρέπεται να έχουμε την ελευθερία κινήσεων μεταξύ κρατών μελών, την οποία έχουμε συνηθίσει και πάνω στην οποία έχουμε οικοδομήσει το σύστημά μας και η οποία έχει πληγεί από την επανεσαγωγή των ελέγχων στα σύνορα που είναι αρνητικές και για τους πολίτες ε, και για την οικονομία. Για να μπορούν λοιπόν όμως να μετακινούνται ελεύθερα οι πολίτες μας θα πρέπει να αναλάβουμε εμείς την ευθύνη αυτή της αναδιοργάνωσης και χαίρομαι που το Κοινοβούλιο μέσω του εισηγητή του κ. Δεμέρα... κατάφερε να πετύχει σημαντική πρόοδο στο θέμα αυτό. Αλλά χρειάζεται κάτι πολύ περισσότερο εάν θέλουμε να αντιμετωπίσουμε με σοβαρό τρόπο τις απειλές κατά των συμπολιτών μας. Χρειαζόμαστε ουσιαστικά ένα ευρωπαϊκό FBI με πλήρεις ε, επιχειρησιακές ικανότητες για να καταπολεμήσουμε το οργανωμένο έγκλημα. Και τι έχουμε στη διάθεσή μας? όχι αυτό που χρειαζόμαστε, που είναι μια ευρωπαϊκή αστυνομία που με δραστήριο τρόπο θα καταπολεμήσει και θα πατάξει αυτές τις εγκληματικές οργανώσεις. Χρειαζόμαστε να περάσουμε πολύ χρόνο ακόμα. Κυρία Κάρη, για ένα λεπτό. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Με τη μεταρρύθμιση της Europol Προχωρούμε σε αστυνομική συνεργασία επί ίσης όρης και με πιο συγκεντρωμένη μορφή που θα μπορούσε να είναι αποτελεσματική ε, στην πάλι κατά του οργανωμένου εγκλήματος. Όμως ε, θα ε, παίρνουμε περισσότερες πληροφορίες για τους πολίτες και το Κοινοβούλιο αυτό νομίζω ότι ελισμόνησε να προστατεύσει αυτή την πτυχή των δεδομένων των προσώπων ε, των, πολιτών. Δηλαδή υπάρχουν ε, δεδομένα στο διαδίκτυο που συλλέγονται και θα πρέπει να δούμε τι είδους δεδομένα συλλέγονται και πώς μπορούμε αποτελεσματικά να τα προστατεύσουμε. Βεβαίως χρειάζεται συνεργασία, προφανώς χρειάζεται ενισχυμένη συνεργασία, αλλά μου φαίνεται ότι πάμε κάπως υπερβολικά μακριά. Ευχαριστώ πολύ κυρία Φεράρα, ένα λεπτό. Ευχαριστώ. Σαν εισηγήτρια της έκθεσης για το οργανωμένο έγκλημα δεν μπορώ παρά να εκφράσω την ικανοποίησή μου για τη συμφωνία αυτή. Είναι πολύ θετικά τα αποτελέσματα τα οποία πετύχαμε στα πλαίσια των διαπραγματεύσεων, έτσι θα κάνουμε την Europol πιο υπεύθυνη και πιο αποτελεσματική ενισχύοντας και τον ελεγκτικό ρόλο των κοινοβουλίων των κρατών μελών, όπως επίσης και τις μορφές προστασίας των προσωπικών δεδομένων. Έτσι η Europol θα ενισχύσει τις προσπάθειες που κάνουν τα κράτη-μέλη στην καταπολέμηση της σοβαρής εγκληματικότητας, θα ενισχύσει τα συστήματα ανταλλαγής πληροφοριών τα οποία δυστυχώς όπως είδαμε δεν έχουν λειτουργήσει μέχρι τώρα. Η καταπολέμηση μαφιόζικου τύπου εγκληματικής δραστηριότητας είναι διαμεθοριακού τύπου και γι' αυτό απαιτείται σε ευρωπαϊκό επίπεδο μια συνολική αντιμετώπιση. Γι' αυτό η δημιουργία κοινών ανακριτικών ομάδων μετά από πρωτοβουλία της Europol και η συνεργασία ανάμεσα στα κράτη-μέλη θα οδηγήσει σε μια νέα περίοδο αποτελεσματικής καταπολέμησης των μαφιόζικων δραστηριοτήτων και της τρομοκρατίας. Ρεμπέγκα, ένα λεπτό. Επίτροπε, συνάδελφοι, ο ρόλος της Europol ήταν η πιο αποτελεσματική συνεργασία ανάμεσα στα κράτη-μέλη σε σχέση με τις ποινικά κολάσιμες δραστηριότητες, φυσικά και εδώ βάζουμε και την τρομοκρατία. Απαιτείται λοιπόν μια δύναμη η οποία να ελέγχει τις ύποπτες δραστηριότητες που θα θέσουν σε κίνδυνο τις ε, ζωές των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Βλέπουμε λοιπόν ότι διευρύνουμε ε, τις αρμοδιότητες της, αλλά δεν της δίνουμε την δυνατότητα ανάληψης πρωτοβουλίας. Πρέπει να ενισχύσουμε την Europol ακόμα περισσότερο. Απαιτείται μια πάρα πολύ ισχυρή υπηρεσία προς το συμφέρον των πολιτών και όχι μια υπηρεσία που να υπόκειται πολιτικά σε άλλα όργανα. Κύριος Κοέγιο ένα λεπτό. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Επίτροπε, αγαπητοί συνάδελφοι, θέλω να συγχαρώ καταρχάς τον κύριο Διάστε Μέρα για την εξαιρετική δουλειά την οποία έκανε μέχρι τώρα. Μας έχει συνηθίσει εμείς θέλουμε μια ενωμένη Ευρώπη η οποία να προστατεύει την ελευθερία των πολιτών της στα πλαίσια του χώρου ελευθερίας δικαιοσύνης. Δεν ανήκουμε σε αυτούς που πιστεύουν ότι είναι αντίθετες μεταξύ τους η ελευθερία και η ασφάλεια. Η ασφάλεια δυστυχώς χωρίς ελευθερία είναι δικτατορία και η ελευθερία χωρίς ασφάλεια είναι η αναρχία. Απαιτείται συνεργασία ανάμεσα στα κράτη-μέλη, ιδιαίτερα σε επίπεδο εσωτερικής ασφάλειας. Η πρόταση που γίνεται είναι πραγματιστική και ισορροπημένη. Είναι κάτι το συγκεκριμένο. Δεν φτιάχνουμε το ευρωπαϊκό FBI. Κάτι τέτοιο δεν θα ήταν δυνατό σε αυτή τη φάση. Είναι όμως μια έκκληση την οποία απευθύνουμε στα κράτη-μέλη. 22 Μαρτίου στις Βρυξέλλες και 13 Νοεμβρίου στο Παρίσι έγιναν απαράδεκτες ε, ε, καταστάσεις οι οποίες έδειξαν ότι οι τρομοκράτες βασίστηκαν στη μη ανταλλαγή ενημερωτικών στοιχείων ανάμεσα στις διάφορες χώρες. Η Ευρώπη λοιπόν έκανε αυτό το οποίο πρέπει. Πρέπει και τα κράτη-μέλη τώρα να συνεργαστούν καλύτερα, να ανταλλάξουν περισσότερες πληροφορίες και να υπάρξει αμοιβαία εμπιστοσύνη, η οποία δεν δημιουργείται με τυχαίο τρόπο. Απαιτούνται μέτρα και ε, συγκεκριμένες συνθήκες. Κύριε Κοέλιο, έχετε μία μπλε κάρτα. Κύριε Βάλτμαντς. Ευχαριστώ. Συμφωνώ με πολλά από αυτά που είπατε για την ελευθερία, την αλληλεγγύη, την υπευθυνότητα. Είπατε όμως ότι η νομοθεσία δεν είναι για ευρωπαϊκό FBI, δεν είναι δυνατόν αυτό. Εμείς θέλαμε να κάνουμε ένα βήμα παραπέρα. Θέλαμε λοιπόν να ρωτήσουμε γιατί δεν είναι δυνατή η ευρωπαϊκή FBI. Εγώ νομίζω ότι χρειάζεται κάτι τέτοιο. Ευχαριστώ πολύ για την ερώτηση αυτή. Ε, Κοιτάξτε, ως ένα βαθμό συμμερίζομαι την άποψή σας, αλλά δεν είναι δυνατόν αυτό τώρα, αυτή τη στιγμή, γιατί αυτό που θέλουμε να κάνουμε είναι να δημιουργήσουμε αμοιβαία εμπιστοσύνη μεταξύ των κρατών μελών. Βλέπουμε σε όλη αυτή τη διαδικασία ότι υπάρχει έλλειψη διαβίβαση δεδομένων γιατί δεν εμπιστεύεται το ένα κράτος μέλος στο άλλο. Να είμαστε ρεαλιστές λοιπόν και λογικοί δεν γίνεται τώρα. Πάμε όσο περισσότερο μακριά μπορούμε. Ε, αυτό, μπορέσαμε να, να, να, αυτό μπορέσαμε να κάνουμε. Κυρία Κινίτσι, πρόεδρε, επίτροπε, θέλω να ευχαριστήσω τον συνάδελφο και όσους συνεργάστηκαν μαζί του για την εξαιρετική προσπάθεια. Η ενημέρωση του διακανονιστικού πλαισίου λειτουργίας της Europol ήταν απαραίτητη για να υπάρξει σωστή συνεργασία ανάμεσα στις αρχές που καταπολεμούν την τρομοκρατία. Τα τελευταία χρόνια η Europol βοήθησε στην καταπολέμηση του διασυνοριακού εγκλήματος δίδοντας ανάλυση, στοιχεία και λειτουργική βοήθεια σε κοινέ δράσεις. Θα πρέπει λοιπόν να λάβουμε υπόψη μας ότι οι νέες απειλές για την ασφάλεια της Ευρώπης απαιτούν μια κοινή απάντηση μετά από τις φαγές των Παρισίων και των Βρυξελών πρέπει να ενισχύσουμε τα μέσα συνεργασίας των, δυνάμεων, των αστυνομικών δυνάμεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρέπει να υπάρχει μια νέα νομική βάση για τη λειτουργία της Europol, για τις νέες αρμοδιότητές της, με σεβασμό στα θεμελιώδη δικαιώματα ο μηχανισμός ελέγχου της λειτουργίας της Europol από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα Κοινοβούλια των κρατών μελών είναι κάτι τον θετικό. Έτσι θα μπορέσουμε να προστατεύσουμε και τα προσωπικά στοιχεία μέσω της πρόβλεψης δημιουργίας μιας υπηρεσίας που θα ελέγχει τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίζεται η Europol τα στοιχεία αυτά σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Τα αποτελέσματα αυτά είναι καρπός τριών χρόνων διαπραγμάτευσης. Πάντως ενισχύεται ο ρόλος της Europol. Πρέπει όμως να υπογραμμίσουμε ότι μόνο η πραγματική συνεργασία ανάμεσα στα κράτη-μέλη θα επιτρέψει στην Europol να λειτουργήσει πιο αποτελεσματικά για να καταπολεμηθεί η διεθνή τρομοκρατία και να στηρίξει τις προσπάθειες εντοπισμού και διάλυσης των τρομοκρατικών δικτύων και σε άλλους τομείς όπως το τράφικινγκ. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Σήμερα μιλάμε για τη Europol. Έχουμε κλασική περίπτωση εδώ στάθμιση συμφερόντων. Από τη μια θέλουμε ενίσχυση της εσωτερικής ασφάλειας, παράλληλα όμως Θέλουμε να δοθεί προτεραιότητα, όσο γίνεται μεγαλύτερη, στην προστασία των δεδομένων. Δηλαδή θα πρέπει να είμαστε πολύ επιλεκτικοί στην ε, συλλογή και διαβίβαση δεδομένων. Αλλά με εξέπληξε το γεγονός ότι κάποιοι ομιλητές επικεντρώθηκαν μόνο στην προστασία δεδομένων και αυτό είναι ελληματικό γιατί η στάθμιση συμφερόντων τι σημαίνει, σημαίνει ότι και τα δύο θα πρέπει να τα σταθμίσουμε. Νομίζω ότι στο σχέδιο αυτό που διαβολευόμαστε ε, δεν καταφέραμε να κάνουμε σωστή στάθμιση συμφερόντων. Θα πρέπει οι υπηρεσίες ασφαλείας να έχουν τα κατάλληλα δεδομένα, τα απαραίτητα και νομίζω ότι αυτό είναι ένα βήμα στη σωστή κατεύθυνση εδώ για να μπορούμε να καταπολεμήσουμε το διασυνοριακό έγκλημα γιατί και με την προσφυγική κρίση είδαμε ότι ιδιαίτερα στη Γερμανία ότι εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι βρίσκονται χωρίς ε, ε, ε, στοιχεία και δεν ξέρουμε από πού προέρχονται. αυτό πρέπει να ληφθεί υπόψη. Ευχαριστώ. Κύριε Κέλμελ, θέλετε να απαντήσετε σε μία μπλε κάρτα από τον κύριο Σάνιν.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 θα χρειαστεί να ξαναξεκινήσετε. Είχαμε κάποιο πρόβλημα ε, σύνδεσης και δεν είχαμε διερμηνία. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να ξανακάνω λοιπόν την ερώτηση. Βλέπετε ότι υπάρχουν τα απαραίτητα εχέγγυα τα οποία θα βοηθήσουν έτσι ώστε κάποια κράτη-μέλη να μην χρησιμοποιήσουν αυτές τις πληροφορίες με τρόπο ο οποίος θα παραβιάσει τα δικαιώματα των ίδιων των πολιτών τους. Ευχαριστώ πολύ για την ερώτηση. Νομίζω ότι δεν μπορούμε να προχωρήσουμε τόσο πολύ στην προστασία δεδομένων να θέτουμε πάντοτε εγγυήσεις αν πάει κάτι στραβά. Ε, υπάρχουν πολλές εκπλήξεις στη ζωή, γι' αυτό μίλησα για στάθμιση συμφερόντων και με αυτόν τον κανονισμό νομίζω ότι θα προς τη σωστή κατεύθυνση. Θα τα θα πρέπει να παρακολουθούμε τις εξελίξεις ε, στην πράξη και θα δούμε αν γίνεται σωστή χρήση των δεδομένων. Εγώ νομίζω ότι θα πρέπει να γίνεται ε, συγκεκριμένη και διαρκής παρακολούθηση. Ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Ρουίς, για ένα λεπτό. Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα σας. Θα ήθελα καταρχήν να συγχαρώ τον εισηγητή, όπως επίσης και τους Σκιώδης, και να σας πω πως οι επαγγελματικές αστυνομίες των δημοκρατικών κρατών αποτελούν έναν πυλώνα για να μπορούμε να ζούμε με ασφάλεια και με πολιτική ελευθερία. Παίζουν τη ζωή τους για μας. Σε μια παγκοσμιοποιημένη χώρα η ενίσχυση της Europol είναι καλό νέο. Γιατί, εάν, ε, γιατί, αυτό, γιατί βέβαια οι κυβερνήσεις θα περιορίσουν τις δυνατότητες παραβίασης που έχει αυτή η υπηρεσία. Έτσι ώστε να έχουμε ε, την κατάλληλη εποπτεία ανθρώπων στο Συμβούλιο που δεν θα είναι ούτε γραφειοκράτες, ούτε ε, άνθρωποι οι οποίοι δεν θα λογοδοτήσουν όταν τους καλέσουμε. Αυτό το οφείλουμε σε όσους ήταν θύματα μέχρι σήμερα εγκληματικών πράξεων και σε όλους τους πολίτες μας. Ε, Πιμέντα Λόπες για ένα λεπτό. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω κυρία Πρόεδρε και να σας πω πως η Europol είναι μια από τις υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που δημιουργήθηκε εδώ και πάρα πολλά χρόνια και στόχος βασικός της Europol είναι η συμμόρφωση με τον νόμο, η επιβολή του νόμου και με τον τρόπο αυτό διευρύνουμε την, ε, το πεδίο ε, και σε άλλες πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης και με τον τρόπο αυτό γινόμαστε πιο παρεμβατικοί. Και τι κάνουμε, περιορίζουμε τις πολιτικές ελευθερίες. Είναι μια δομή την οποία επιβάλλουμε στα κράτη-μέλη κατά της εθνικής ε, κυριαρχίας και κατά της αυτονομίας των εθνικών διοκτικών αρχών. Επιβάλλουμε μια αναπόφευκτη συνεργασία μέσω μηχανισμών και δομών που υπάρχουν. Θα μπορούσαμε να έχουμε καταφέρει κάτι αντίστοιχο χωρίς ε, να κάνουμε αυτό που προτείνεται εδώ, που είναι ένας περιορισμός των θεμελιωδών δικαιωμάτων των συμπολιτών μας. Εμείς ε, βεβαίως είμαστε κατά. Κύριο Ζεντεχόφσκι, ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε. Ε, δεν συμφωνώ με τον ε, ομιλητή. Καμιά φορά δεν έχει νόημα και γενικά άκουσα πολλές παρεμβάσεις που δείχνουν ότι οι ομιλητές δεν διάβασαν το κείμενο και δεν έχουν ιδέα τι κάνει η Europol. Προσωπικά θεωρώ ότι η Europol είναι από του σημαντικότερους οργανισμούς, ε, ένα σημαντικό μέσο για την ασφάλεια στην Ευρώπη. Τα προηγούμενα χρόνια ε, πίστηκα ότι ε, υπάρχουν αδυναμίες και ελλείψεις στο έργο που επιτελεί και αυτό προσπαθούμε να διορθώσουμε εδώ. οι ανώτεροι υπάλληλοι και η Europol θα πρέπει να προβαίνουν σε αμοιβαία ανταλλαγή πληροφοριών για δυνητικά επικίνδυνα πρόσωπα. Αλλιώς πώς θα καταπολεμηθεί το οργανωμένο έγκλημα ή η τρομοκρατία, πώς θα δράσουν για την ασφάλεια των πολιτών της Ευρώπης. Στη σημερινή Ευρώπη ε, τα προβλήματα είναι πολλά και χρειάζεται καλύτερο συντονισμός. Γι' αυτό νομίζω ότι μακροπρόθεσμα πρέπει να ενισχυθεί η Europol, όχι μόνο οικονομικά, αλλά και στις αρμοδιότητές της. Αυτό δεν γίνεται βέβαια χωρίς αναδιοργάνωση της συνεργασίας μεταξύ των διαφορετικών εθνικών και ευρωπαϊκών αρχών. Κανένας οργανισμός δεν μπορεί να αντιδράσει στις νέες προκλήσεις με ευέλικτο τρόπο αν δεν διαθέτει η ίδια αρκετή ευελιξία. Χρειάζεται λοιπόν ε, αύξηση οικονομικών και ανθρώπινων πόρων. Ευχαριστώ. Ο κύριος ε, κυρία Τόμασιτς. Ευχαριστώ πολύ. Ε, στηρίζω αυτή την νομοθετική πρωτοβουλία γιατί δίνει νέες αρμοδιότητες στην Europol, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά επιμόρφωση και μετεκπαίδευση των αστυνομικών, χωρίς να υπησέρχεται στην ε, ε, κυριαρχία των κρατών μελών. Δεν πειράζει την επικουρικότητα. Πιστεύω ότι η λύση ότι κάθε κράτος μέλος θα πρέπει να έχει μια ειδική μονάδα ως σύνδεσμο μεταξύ Europol και εθνικών αρχών πιστεύω ότι είναι πάρα πολύ κατάλληλη η λύση αυτή διότι θα διατηρήσει τις αρμοδιότητες των κρατών μελών χωρίς να επηρεάσει αρνητικά τις αρμοδιότητες της Europol. Χρειάζεται και ενισχυμένος έλεγχος στην Europol. Ε, αυτό θα το αναλάβουν το Ευρωπαϊκό και τα Εθνικά Κοινοβούλια ε, για να υπάρχει διαφάνεια και προ, ε, σεβασμός των δεδομένων το διαδίκτυο ε, ε, βοήθησε τις δραστηριότητες των εγκληματικών ε, οργανώσεων και γι' αυτό ακριβώς χρειάζεται δράση της Europol και σε αυτό το επίπεδο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Η Ευρώπη μπορεί να εξοπλιστεί καλύτερα ε, τώρα και να καταπολεμήσει αποτελεσματικότερα το οργανωμένο έγκλημα. Ε, αντιδρούμε ταχύτερα σε έναν κόσμο που γίνεται μικρότερος. Είναι σημαντικό να έχει ε, ενισχυμένη εντολή η Europol για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και του οργανωμένου εγκλήματος. Αυτό είναι εκ των ονουκάνευ. Θα πρέπει να μπορούμε να αντιδρούμε γρήγορα και να καταπολεμούμε τα αδικήματα αυτά. Για πολλά χρόνια και στην επαγγελματική μου σταδιοδρομία, στην αστυνομία, είδα ότι η εγκληματικότητα γίνεται, διεθνοποιείται όλο και περισσότερο και πρέπει και εμείς να ε, παρεμβαίνουμε με αποτελεσματικότερο και ταχύτερο τρόπο δεν ε, ε, πρόκειται μόνο για αυτό που ανέφερε η κυρία Χολμάιερ. Θέλουμε ε, πολύ σημαντική συνεργασία και γι' αυτό θα φροντίσουμε. Ευχαριστώ πολύ. Κυρία Πρόεδρε, κυρία Επίτροπε, είναι καλή ημέρα αυτή διότι ε, είναι επικοδομητική η πλειοψηφία αυτού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου υπέρ τη ενίσχυσης της Europol. Συγχαρητήρια στον εισηγητή, ο οποίος ε, όλα τα προηγούμενα χρόνια συνεργάστηκε με τους Σκιώδης. Θα ήθελα να αναφερθώ στην επόμενη φάση της ε, εξέλιξης όμως. Χαιρετίζω την ανακοίνωση του Επιτρόπου Αβραμόπουλου για την ενίσχυση της Europol σε επόμενα στάδια, κατά την επόμενη διετία, ούτως ώστε να αντιμετωπίσουμε ε, τις νέες ανάγκες στην πάλη ε, κατά του οργανωμένου εγκλήματος και της τρομοκρατίας. Ε, με βάση το, τη σημερινή σύνθεση της Europol είναι σαφές ότι ο συντονισμός και η συνεργασία δεν μπορούν να έχουν πλήρη επιτυχία ε, στην καταπολέμηση της τρομοκρατίας και του οργανωμένου εγκλήματος. Η Ευρώπη πρέπει λοιπόν να κερδίσει αυτή την τρομερή μάχη. Άρα πρέπει να είναι πιο ενισχυμένη η Ευρώπη. Άρα ε, θα πρέπει να υπάρξει μια Ευρωπαϊκή Ένωση Ασφάλειας όπου η Europol θα είναι ε, μια υπερεθνική μονάδα με κεντρική διοίκηση και θα μπορεί να παρεμβαίνει διασυνοριακά σε ολόκληρη την Ευρώπη. Ε, αυτό είναι ένα μεγάλο επόμενο βήμα και εύχομαι να ανταποκριθεί σε αυτό και να εργαστεί αποτελεσματικά η Κομισιόν. Ευρωπαϊκό FBI μπορεί να δημιουργηθεί στην, ε, στο τέλος σε μια Ευρωπαϊκή Ένωση η οποία θα είναι στιβαρή και θα μπορεί να εγγυάται την προστασία των πολιτών της. Ευχαριστώ. Κύριος Νομίζω ότι μπορώ να πω χωρίς να διαψευστώ ότι η Europol με μεγάλη επαγγελματικότητα και με θετικά αποτελέσματα φέρει εις πέρα στην αποστολή της. Αλλά το διεθνές σκηνικό έχει αλλάξει. Τα πράγματα αλλάζουν με πολύ μεγάλη ταχύτητα. Βλέπουμε τι έγινε στο Παρίσι και στις Βεξέλες. Βλέπουμε τι γίνεται με τη μετανάστευση και γι' αυτό σήμερα περισσότερο από ότι στο παρελθόν απαιτείται ενίσχυση της Europol αύξηση των πιστώσεων για τη λειτουργία της, αύξηση του οργανογράμματος, αύξηση των μέσων, έτσι ώστε με ευφυή τρόπο να δοθεί η δυνατότητα ε, καταπολέμησης της ε, ηλεκτρονικής εγκληματικότητας και των τρομοκρατικών προσπαθειών στο διαδίκτυο. Απαιτείται νέα μορφή συλλογή πληροφοριών από τα κράτη-μέλη και συνεργασία και γι' αυτό ακριβώς η πρόταση νομίζω ότι είναι πολύ θετική. Ο κύριος Ράγγελ, 1,5 λεπτό. Ευχαριστώ, πολύ. Θα ήθελα καταρχήν να συγχαρώ τον συνάδελφο κύριο Δίας. Έκανε πολύ καλή δουλειά. Πραγματικά είναι καταπληκτική η γνωμοδότηση αυτή, η έκθεση μάλλον, και θα ήθελα ως μέτρο της, ε, ως μέλος της ε, Επιτροπής Συνταγματικών Θεμάτων να αναφερθώ σε αυτήν την ουσιαστική αναθεώρηση ε, του κανονισμού της Europol και να σας πω πως πρώτα απ' όλα προσαρμόζουμε την Ευρωπόλ στη συνθήκη της Λισαβόνας, κάτι το οποίο ήταν εξαιρετικά σημαντικό. Και σε επίπεδο κοινοβουλευτικού ελέγχου νομίζω πως δημιουργούμε εδώ ένα στοιχείο κλειδί γιατί θα πρέπει να υπάρχει λογοδοσία από το όργανο αυτό προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Επίσης έχουμε μια σειρά από εχέγγυα για την προστασία δεδομένων, για τη μάχη κατά του καταπολ κατά του οργανωμένου εγκλήματο όπου χρειάζεται συντονισμό και ανταλλαγή ή πληροφοριών οι οποίε πολλές φορές είναι ευαίσθητε. Και νομίζω πως θα πρέπει ο έλεγχο και η υποπτία αυτής τη πτυχή να γίνεται με τον ενδεδειγμένο τρόπο. Θα ήθελα να τονίσω και να σταθώ σε ένα σημείο ακόμα. Μιλάμε για διεθνέ έγκλημα, έγκλημα χωρί σύνορα. Ε, δεν είναι κάτι άγνωστο αυτό, είναι κάτι το οποίο είχαμε εδώ και χρόνια. Το έγκλημα εδώ και δεκαετίες έχει οργανωθεί σε δίκτυα διεθνή, άρα λοιπόν θα πρέπει να δημιουργήσουμε και στα δικά μας δίκτυα για να τα καταπολεμήσουμε. Και νομίζω ότι κάνουμε ένα πολύ καλό βήμα για να οργανώσουμε ένα αστυνομικό σώμα το οποίο θα μπορεί να αντιμετωπίσει με μεγαλύτερη ευκολία αυτό το οργανωμένο έγκλημα. Θα περάσουμε λοιπόν στο Catch the Eye. Η κυρία Αγιάλα Σέντερ είναι η πρώτη μας ομιλήτρια. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω καταρχήν τον κύριο Δίας Δεμέρα και τους υπόλοιπους συναδέλφους ε, για ε, τον τρόπο με τον οποίο αντιμετώπισαν το θέμα αυτό και μας βοήθησαν να προχωρήσουμε στο κανονισμό αυτό. Οι τελευταίες επιθέσεις στις Βρυξέλλες και στο Παρίσι, αλλά επίσης και στο Λονδίνο και στην Μαδρίτη έδειξαν πως επήγε να έχουμε το ε, συνενετικό και στέρεο νομικό πλαίσιο το οποίο θα επιτρέψει στις δικές μας διοκτικές αρχές να συνεργαστούν, να στηριχθούν από τη Europol για να τα πάνε καλύτερα. Ο κανονισμός αυτός σημαίνει μεγαλύτερη επένδυση στην πρόληψη, στην ανάλυση κινδύνου, στη συνεργασία και περισσότερες ε, μυστικές πληροφορίες που θα ανταλλάσσονται με ε, τους μυστικούς πράκτορες που θα μας επιτρέψουν να παρακολουθήσουμε από μέσα τι γίνεται. Όχι μόνο για την τρομοκρατία αλλά και για άλλες εγκληματικότητες που είναι ε, το τράφικο, το, το τράφικο με συγχωρείτε, το ξέπλυμα ε, όπως επίσης και οι κυβερνοεπιθέσεις σε κοινωνίες όπως οι δικές μας. Σας ευχαριστώ πολύ. Τα χρόνια διαρκώς αυξάνονται τόσο οι δυνατότητες όσο και ο προπολογισμό της Europol, ειδικά στον τομέα της καταπολέμησης της τρομοκρατίας. Τα πρακτικά αποτελέσματα όμως είναι απογοητευτικά. Αυτό άλλωστε φάνηκε πρόσφατα τόσο στη Γαλλία όσο και στο Βέλγιο οπωσδήποτε πρέπει να δοθεί έμφαση στην καταπολέμηση της τρομοκρατίας ιδιαίτερα σε συγκεκριμένες περιοχές κρατών μελών. αυτό όμως πρέπει να γίνει με σεβασμό στον ιδιωτικό βίο των πολιτών της ένωσης. αντίθετα επιχειρείται στο όνομα της καταπολέμησης της τρομοκρατίας να τροφοδοτηθεί από τους κρατικούς προϋπολογισμούς η περαιτέρω καταστολή και επιτήρηση των πολιτών σε πανευρωπαϊκό επίπεδο και ενώ αποδεδειγμένα αυτή η πολιτική έχει δείξει τα όρια της στην καταπολέμηση της τρομοκρατίας η ευρωπαϊκή ένωση οφείλει να ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να δαπανίσουν χρήματα στη φύλαξη των συνόρων τους καθώς επίσης και σε προγράμματα κοινωνικής ένταξης και απασχόλησης των μουσουλμανικών πληθυσμών που ζουν επί δεκαετίες σε κράτη μέλη της ευρωπαϊκής ένωσης. αυτός είναι ο μοναδικός δρόμος για μια αποτελεσματική πρόληψη του φαινομένου της τρομοκρατίας. ευχαριστώ. Θα δώσω το λόγο στον κύριο Καπούτο, αλλά τον παρακαλώ να μην μιλάει πάρα πολύ γρήγορα. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Οι πρόσφατες τρομοκρατικές ενέργειες και η παρουσία των τρομοκρατικών ομάδων στο διαδίκτυο απαιτεί καλύτερη συλλογή πληροφοριών και κοινή δράση περισσότερες εξουσίες στην Ευρωπολ δυνατότητα άμεσης καταπολέμησης των τρομοκρατικών απειλών και ιδιαίτερα ο ρόλος ε, του Internet Referral Unit που θα καταπολεμήσει την online προπαγάνδα των τρομοκρατών θα πρέπει να στηρίξει ε, τις προσπάθειες των κρατών μελών. Οι νέοι κανόνες λειτουργίας θα ενισχύσουν τις δυνατότητες της Europol να καταπολεμήσει την τρομοκρατία και την ε, εγκληματικότητα τη δικτυακή. Έχουν λοιπόν βήματα προς τα εμπρός, δεν είναι επαρκή Μιας και είναι πάντα υψηλό το επίπεδο της απειλής, απαιτείται περαιτέρω ενίσχυση της Europol και για τις ενέργειες τις οποίες κάνει στο πεδίο και για τις ανταλλαγές πληροφοριών σε σχέση με εγκληματικές δραστηριότητες. Ο κύριος Γιάκοφτσιτς. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ. Στην Ευρώπη χρειαζόμαστε μια ένωση ενημέρωσης και ειδήσεων σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι δεν, υπάρχουν, δεν γίνονται συμβιβασμοί με τους εγκληματίες. Γι' αυτό χρειάζεται ένα βήμα παραπέρα, το ταχύτερο δυνατόν μάλιστα. Καταλαβαίνω ότι στους κόλπους της Ένωσης υπάρχουν διαφορετικές απόψεις όταν πρόκειται για την αντίδραση σε επιθέσεις. Αλλά όταν αντιμετωπίζουμε την τρομοκρατία ε, πρέπει να είμαστε ενωμένοι. Είδαμε τι έγινε τους τελευταίους μήνες. Υπάρχουν ε, απειλές ε, και βέβαια αναγκαστήκαμε να περιορίσουμε την ελεύθερη διακίνηση. Χρειάζεται ανταλλαγή πληροφοριών κατεπηγόντως και να καλύπτει πολλές πληροφορίες. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Οι Ευρωπαίοι πολίτες χρειάζονται ένα καλύτερο νομικό πλαίσιο για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας. Απαιτείται καλύτερη συνεργασία διασυνοριακή. Είναι ένα από τα νομοθετικά κείμενα τα οποία θα έλεγα ενδιαφέρουν ιδιαίτερα και δίνουν την δυνατότητα παρέμβασης και ελέγχου και στα κοινοβούλια των κρατών μελών και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Η προστασία των προσωπικών δεδομένων είναι καθοριστική, αλλά αυτό δεν θα πρέπει όμως να θέτει σε κίνδυνο την ασφάλεια. Η βελτίωση λοιπόν της Europol θα προσδώσει περισσότερη ασφάλεια στους πολίτες της Ένωσης. Θα πρέπει λοιπόν να μην είναι η αχίλιος πτέρνα ε, ε, της προσπάθειας καταπολέμησης της τρομοκρατίας. Η ανταλλαγή πληροφοριών μέχρι τώρα δεν δούλεψε. Αυτό θα πρέπει να διορθωθεί και δεν θα πρέπει να κάνουμε καμία υποχώρηση προς αυτό. Ο κύριος Αγγιλάρ, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω και να συνταχθώ κι εγώ με όσους αυτή τη στιγμή συγχαίρουν τον ε, εισηγητή για την ολοκλήρωση αυτού του κειμένου, τον κύριο Δίας Μέρα, γιατί πραγματικά η δουλειά που έκανε ήταν να ενημερώσει ε, την νομοθεσία μας, να τη συνδέσει με τη Λισαβόνα και να επιτρέψει μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα στο εργολείο αυτό. Τράφικινγκ, ε, λαθρεμπόριο, όπλο, ναρκωτικών, ε, νομιμοποίηση παράνομου χρήματος. Έτσι λοιπόν έχουμε μία πιο ενημερωμένη Europol που χρειάζεται κάτι ακόμα, την πολιτική βούληση να γίνει η Europol μια εμβριακή μορφή του ευρωπαϊκού FBI που τόσο βοήθησε ε, στη μάχη ε, κατά του εγκλήματος και της ασφάλειας της ΕΠΑ και είναι κάτι απαραίτητο για να μην υπάρχει πια ατιμορρησία ακριβώς επειδή κάποιος πέρασε από το ένα σύνορο στο άλλο. Θα πρέπει να διδαχθούμε εμείς οι Ευρωπαίοι από το FBI και να κάνουμε κάτι αντίστοιχο στην Ευρώπη. Η κυρία ε, Φλασίκοβα, επόμενη μιλήτρια. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε, κυρία Επίτροπε. Χαιρετίζω την ε, μεταρρύθμιση αυτή των διοκτικών αρχών μετά από τα τρομοκρατικά πλήγματα Πρέπει η Europol να δρά αποτελεσματικότερα και ταχύτερα στις τρομοκρατικές απειλές και η ασφάλεια των πολιτών πρέπει να είναι στην πρώτη γραμμή. Άρα λοιπόν χρειάζεται εντατικότερη συνεργασία και έλεγχος ε, πριν ε, ως πρόληψη των αδικημάτων. Όλα αυτά θα πρέπει να τα διασφαλίσουμε. Οι ερευνητές, οι έρευνες στην Europol πρέπει να γίνονται και διασυνοριακά. Γι' αυτό χρειάζονται πόροι. Ε, οι ελευθερίες των πολιτών μας δεν θα περιοριστούν, αντίθετα θα προστατευτούν. Ε, θα, έτσι κι αλλιώς η Europol θα υπόκειται στο δημοκρατικό έλεγχο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των Εθνικών Κοινοβουλίων. Ευχαριστώ. Ο κύριος Αβραμόπουλος έχει το λόγο για να κλείσει τη συζήτηση, μια και τελείωσε και η διαδικασία Catch the Eye. Ευχαριστώ πολύ. Αξιότιμα μέλη, καταρχήν να ευχαριστήσω για τη συμβολή στη συζήτηση. Ο κοινός παρονομαστής ε, όλων των ε, παρεμβάσεων είναι ότι πρέπει να αντιδράσουμε στην ανάγκη των πολιτών για μεγαλύτερη ασφάλεια. Και αυτό προσπαθούμε να κάνουμε με αυτή τη μεταρρύθμιση. Όλοι γνωρίζουμε ότι η τρομοκρατία και το σοβαρό υπερεθνικό έγκλημα, όπως είπατε και συμφωνώ και εγώ, δεν γνωρίζει σύνορα. Οι δικές μας ιδιοκτικές αρχές, αρμόδιες για την επιβολή του νόμου, είναι και αρμόδιες για την ασφάλεια των πολιτών μας. Για να μπορέσουμε να εντοπίσουμε αποτελεσματικά τους δράστες, χρειάζεται ένα κέντρο ανταλλαγής πληροφοριών με πλήρη επιχειρησιακή και αναλυτική υποστήριξη. Με το βελτιωμένο πλαίσιο που δημιουργούμε, η Europol θα μπορεί να ε, δρά συνδυαστικά και να δίνει στα κράτη-μέλη την υποστήριξη που χρειάζεται για να καταπολεμήσουν την τρομοκρατία και το σοβαρό έγκλημα. Η Ευρώπη θα μπορέσει να το κάνει αυτό πιο αποτελεσματικά και πιο αποδοτικά τώρα θα είναι πιο υπόλογη και θα εργαστεί ε, με πλήρη σεβασμό των κανόνων προστασίας δεδομένων. Σας ενθαρρύνω σήμερα και σας καλώ να ψηφίσετε υπέρ του συμβιβαστικού κειμένου το οποίο ε, θέτει σε εφαρμογή αυτά που συζητούσαμε για χρόνια. Ας φροντίσουμε ούτω ώστε να λειτουργήσει υπέρ των πολιτών της Ένωσής μας. Ευχαριστώ. Κύριε Διαζεμέρα, θέλετε να κλείσετε κι εσείς. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω και τον κύριο Αβραμόπουλο. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω και για τις δύο παρεμβάσεις που κάνατε και πραγματικά εκτιμώ τα λόγια σας γιατί πραγματικά κύριε Αβραμόπουλε ε, θίξατε ακριβώς τον πυρήνα του θέματος. Χρειάζεται περισσότερος κοινοβουλευτικός έλεγχος, μεγαλύτερη ανάλυση δεδομένων, περισσότερη ανταλλαγή και προστασία προσωπικών δεδομένων. Χρειαζόμαστε μια υπηρεσία η οποία θα αποτελεί έναν ισχυρό κόμβο ανταλλαγής πληροφοριών και όπου θα έχει αναπτυγμένες αναλυτικές δυνατότητες για να προστατεύει τους Ευρωπαίους. Ένα μόνο σημείο Στηρίζω τα όσα είπε η συνάδελφος Μάιτε για την διακυβέρνηση. Θα πρέπει το Συμβούλιο ε, αυτό της Europol να είναι επαγγελματίες και όχι πολιτικοί. Και για τα όσα είπαν οι συνάδελφοι, τους ευχαριστώ ιδιαίτερα. Και θα κάνω μία περίληψη. 42 παρεμβάσεις έγιναν. Κάποιες βασίστηκαν στην γνώση του αντικειμένου, άλλες βασίστηκαν στην ε, κατανόηση ε, του ε, αντικειμένου συναισθηματικά. Όλες είναι αξιοσέβαστες. Θα ήθελα να ευχαριστήσω πάρα πολύ όσους συμπίτουν και να λυπηθώ για όσους έχουν αντιρρήσει το τι κάνουμε, αλλά αποτελεί αυτό αναφέρεται το δικαίωμά τους. Και να σας πω πως από τις 42 παρεμβάσεις, 32 στήριξαν τον εισηγητή και έξι που ζητούν μια πιο ισχυρή Europol και αυτή είναι κυρίως φιλελεύθερη και θα ήθελα να κλείσω απευθυνόμενος τους πράσινους και να τους πω πως βεβαίως εκτιμώ την πολιτική σας ε, στήριξη ε, και την δική σας πολιτική συστράτευση. Ο κανονισμός ε, Europol ε, καταλαβαίνω ότι χρειάστηκε από την πλευρά σας να υποβληθεί και μία ε, τροπολογία που είναι περισσότερο ε, μορφής και όχι τόσο ουσίας γιατί έχει να κάνει με τον τρόπο το οποίο θα διατυπώνουμε τις διαδικασίες για το IRU. Σας ευχαριστώ όλους για τα καλά σας λόγια. Σας ευχαριστώ πολύ.